do Okay, let's do robotics. Ας πάμε στη ρομποτική λοιπόν. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα με την πολύ αναμενόμενη αυτή γνωμοδότηση. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Υπάρχει εδώ συνάδελφος από την Κομισιόν. Όχι, αλλά θα ξεκινήσουμε ούτως ή άλλως. Λοιπόν, είμαστε στο σημείο 5, συνάδελφοι. Σχέδιο γνωμοδότησης του κυρίου Μπένι με την έκθεση ίδια πρωτοβουλία για την ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική, όπω γνωρίζουν οι συνάδελφοι. Είναι συνδεδεμένη η Επιτροπή, η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ στι οθόνε. Έχουμε ψηφοφορία. Τέλο πάντων, συνεχίζω. Ε, συνδεόμαστε δυνάμει του, του άρθρου 54 για αυτό το θέμα, αλλά φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική είναι κάτι στο οποίο έχουμε και εμείς να δώσουμε μια καθοριστική γνωμοδότηση, όπως και για άλλα. Στις 23 Οκτωβρίου συμφώνησαν λοιπόν οι συντονιστές ότι λόγω των στενών χρονικών περιθωριών ε, η γνωμοδότηση θα συντασσόταν ε, από τη Λίμπε μόνο στα αγγλικά, αλλά είναι σημαντικό το θέμα, οπότε να ζητήσω από τον κύριο Μπόνη να μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησης και μετά θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποια συζήτηση. Μίχαλ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε όλοι, η τεχνητή νοημοσύνη είναι μία από τις ε, τεχνολογικές στρατηγικές ε, του 20 ου προδεώνα παγκοσμίω και για την Ευρώπη. Θα επιφέρει θετικές ε, μεταβολές στην ευρωπαϊκή οικονομία όσον αφορά την καινοτομία, την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα την ευημερία των πολιτών μας. Θα μας βοηθήσει να βελτιστοποιήσουμε την παραγωγή, να ε, χρησιμοποιήσουμε στοιχεία προβλέψεων σε πολλούς πολλούς τομείς και προγνώσεις. Από την άλλη όμως αποτελεί κάποιο είδους μάχη μεταξύ ζωφερών ε, και αισιόδοξων σενάριων. Μιλάμε για την υγεία με τα προηγμένα συστήματα τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα στις ε, υπηρεσίες ε, πρώτης βοήθειας να διαγνώσουν καρδιακές, καρδιακά προβλήματα απειλητικά για την υγεία ή άλλες απειλητικές καταστάσεις σε όλα αυτά τα θέματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά θα μπορούσε κανεί να μιλήσει για αισιόδοξα ωφέλη. Αλλά όπω το βλέπουμε εμεί, υπάρχουν και κάποιε απειλέ για την ε, αγορά εργασία από την τεχνητή νοημοσύνη. Η ταχεία λοιπόν εξέλιξη των νέων τεχνολογιών τη τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί και συνεπάγεται και κάποιε απειλέ. Διότι η κακόβουλη χρήση τη τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να απειλήσει πρώτα απ' όλα την ψηφιακή ασφάλεια μέσω μηχανημάτων ε, εκπαίδευσης εγκληματιών που θα πλήξουν τη φυσική ασφαλεία ε, και μάλιστα εδώ μιλάμε για έξω ε, κυβερνητικούς παράγοντες που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για κλιματικές δραστηριότητες, για διακίνηση ναρκωτικών, για την πολιτική ασφάλεια, για το profiling, για την καταστολή και για εκστρατείες παραπληροφόρησης. Η τεχνητή νοημοσύνη πράγματι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή ευρεία ε, κλίμακας ε, επιθέσεων ε, πολύ αποτελεσματικών. Το Κοινοβούλιο λοιπόν θα πρέπει να πραγματοποιήσει ολιστική ανθρωποκεντρική προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη της στρατηγικής τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό. στη Γαλλία, στη Γερμανία, στη Φιλανδία, στην Εστονία και στην Πολωνία ε, πολλοί παραγωγοί λένε ότι θέλουν τις δικές τους στρατηγικές αλλά πρέπει να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό διότι θα αποτελέσει πλεονέκτημα εμπορικό για μας και κοινωνικό να έχουμε μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση όπου τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη-μέλη και τα ερευνητικά κέντρα θα συνεργάζονται για μια κοινή προσέγγιση. Αναμφίβολα η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως ε, θεσπίζεται στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ειδικότερα θα πρέπει να συμμορφώνεται με την προστασία των δεδομένων, το ιδιωτικό απόρριτο και την ασφάλεια καθώς και με τους ε, κανόνες του GDPR. Αυτό ε, είναι ένα από τα σημεία στο οποίο εστιάζομαι στο σχέδιο γνωμοδότησής μου και ε, έτσι θα συμβάλλω στην έκθεση της Επιτροπή Ήτρε με αυτά τα στοιχεία. Στο σχέδιο γνωμοδότησής μου επίσης αναφέρομαι και στα ηθικά ζητήματα που απορρέουν από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης εστιαζόμενος στην διαφάνεια και στην ε, τεκμηρίωση αυτό είναι ένα από τα βασικά ζητήματα για τους αλγόριθμους, όπως και στη δικαιοσύνη και στις ίσες ευκαιρίες. Ε, όπως ξέρετε, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έχει ε, προετοιμάσει μια έκθεση για τους αλγόριθμους και τους κινδύνους της διακριτικής μεταχείρισης. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Πιστεύω ακράδαντα ότι η ανθρώπινη κατανόηση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης είναι κέρια σημασίας ώστε να υπάρξει ευαισθητοποίηση και εμπιστοσύνη μεταξύ των καταναλωτών οι οποίοι με τη σειρά τους ε, θα βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο να προοδεύσει περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη. Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τους. Επίσης θα πρέπει να μπορούν να γνωρίζουν ε, ότι πότε ε, επικοινωνούν ή αλληλεπιδρούν με μηχάνημα και έτσι θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην αλληλεπίδραση με τα συστήματα τεχνητή νοημοσύνη. Πολλέ αναλύσει σήμερα εστιάζονται στη σχέση και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπων και των chatbox, ε, ε, chatbox που βασίζονται στη μηχανική εκμάθηση. Τα chatbox που βασίζονται σε marketing δεν ε, εστιάζονται ως μηχανήματα με δυνατότητα εκμάθησης. Λένε είμαστε άνθρωποι όταν τους ρωτούν άνθρωποι. Οπότε είναι σαφώς ότι χρειαζόμαστε σαφείς ε, κανόνες. Κάτι άλλο σημαντικό, οι δυνατότητες ελέγχου. Διότι η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς αναπτύσσεται, θα πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε από ανθρώπους, ώστε να αποφύγουμε προβλήματα στο μέλλον. Τέλος, στο σχέδιο γνωμοδοτησίσμου μιλάω για τη σπουδαιότητα της ποιότητας των δεδομένων ε, για την αναπτύξη αλγορίθμων, η χρήση χαμηλής ποιότητας απερχαιωμένων δεδομένων, ατελών δεδομένων, μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκείς προβλέψεις που θα οδηγήσουν σε διακριτική μεταχείριση και προκατάληψη. Είναι σημαντικό λοιπόν οι αλγόριθμοι να έχουν διαμορφωθεί βάσει αντιπροσωπευτικών δεδομένων ε, υψηλής ποιότητας, ώστε να υπάρχει στατιστική ισότητα η ανάπτυξη μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ σημαντική. Θα διασφαλίσει ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασία δεδομένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αξιών, ηθικών ζητημάτων θα αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη των ε, συστημάτων ρομποτική και τεχνητής νοημοσύνης. Περιμένω λοιπόν ε, με ανυπομονησία τη συνεργασία μας ε, σε αυτή τη γνωμοδότηση με τους και συζητητέ. Ευχαριστώ. Πράγματι έχετε δίκιο, είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα, ζητήματα ιδιωτικότητος από αυτά που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ, δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό θα πάω στους συναδέλφους απευθείας που θέλουν το λόγο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο ο κύριος Πάντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο επηρεάζει την καθημερινή ζωή μας ε, και την επηρεάζει σημαντική. Είναι σημαντικό στην περιοχή αυτή η Ευρώπη να είναι ηγέτης ώστε να αναπτυχθεί μια τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης επί τη βάση αρχών που να είναι διαφανής. Μία από τις ε, πιο βασικές προκλήσεις προκειμένου να διατηρήσουμε σε αυτό το πεδίο την ανταγωνιστικότητά μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιείται ε, σε ένα ευρύ φάσμα της βιομηχανίας, γιατί αυτή τη στιγμή, ή μάλλον το 2017, το 25 μόνο των επιχειρήσεών μας ε, χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογίες και μεταξύ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μόνο το 10%. Για να ενισχύσουμε τους αριθμούς αυτούς θα πρέπει να ενισχύσουμε και τις επενδύσεις. Αυτό είναι κρίσιμη σημασία, ακόμα πιο κρίσιμο είναι το γεγονό ότι οι οποιασδήποτε εξελίξεις τη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης δεν θα πρέπει να γίνονται ει βάρο των υπολείπων ενδιαφερομένων και των πολιτών. Διότι πλήττεται η εμπιστοσύνη που έχει το κοινό που έχουν οι πολίτες σε αυτές τις τεχνολογίες με μερικά κρούσματα που παρατηρούμε. Η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να βασίζεται, να παρακολουθεί μάλλον, τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων άρθρα 7 και 8 αλλά και ε, κατάλληλες διατάξεις ε, της ε, νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα προστατεύεται λοιπόν η ιδιωτικότητα αλλά από την άλλη να αντιμετωπίσουμε κάποιες ίσως εσφαλμένες και προκατασκευασμένες ιδέες που έχει το κοινό σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας αυτής. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εγώ λέει ο Πρόεδρος. η κυρία Γκόμη. Ε, πρόεδρε, δεν θα μπορούσα παρά να συμφωνήσω απολύτω με τον κύριο Μπόνι ότι εδώ το διακύβευμα είναι η ηθική, μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση καθότι πλέον, λέει η ομιλήτρια, οι μηχανές μπορούν να μαθαίνουν από μόνες τους. Και επίσης, το πρόβλημα είναι να μην μείνουμε πίσω. Αυτά ήδη χρησιμοποιούνται, οι τεχνολογίες αυτές ήδη υφίστανται. Ήδη στην Κίνα έχουν αυτό το credit scoring, αυτό το σύστημα που παρακολουθεί και την συμπεριφορά, αν θέλετε, και τη στάση των πολιτών. Έχουν μια βαθμολόγηση οι πολίτες χρησιμοποιώντα ένα τέτοιο σύστημα. Επίση πρόσφατα έμαθα για μια γερμανική επιχείρηση που φιλοδοξεί να είναι η Amazon της χρηματοδότησης των καταναλωτών και ερευνά τα στοιχεία της προσωπικότητας τα οποία τηρούνται μεταξύ των δεδομένων στην πλατφόρμα της Facebook μεταξύ άλλων. Επίσης ε, χρησιμοποιούνται αντίστοιχα δεδομένα για την ε, δανειοδότηση σε χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Δηλαδή, πώς θα εξασφαλίσουμε ότι αυτού του είδους οι θεμελιώδεις ανησυχίες θα γίνουν σεβαστές και θα καλυφθούν σε σχέση με μηχανήματα που θα χρησιμοποιούμε καθημερινά στη ζωή μας. Γιατί όπως είπε και ο κύριος Μπόνι, δεν αναφερόμαστε μόνο σε μηχανήματα περιθωριακά, αλλά καθημερινή χρήση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος η Κομισιόν. Έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μας δίνετε το λόγο. Συμφωνούμε πράγματι ότι πρέπει να είναι κανείς εξαιρετικά προσεκτικός ζυγίζοντας και τις ωφέλειες αλλά και την δυνητική απειλή. Αυτό είναι μέρος της στρατηγικής μας ώστε να έχουμε μια συνολική προσέγγιση στο ζήτημα. Και εδώ θα πρέπει να διαβολευτούμε και με τους ερευνητές της τεχνολογίας, το οποίο και πράττουμε στα πλαίσια των ε, συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα, για παράδειγμα στην χρηματοδότηση των προγραμμάτων του ορίζοντα 2020 αλλά και γενικώ όλων των προγραμμάτων μας. Όμως το θέμα είναι διατομεακό στη φύση του. Δεν είναι μόνο τεχνολογικής φύσεως το ζήτημα αλλά κοινωνικής, νομικής, ηθικής κτλ. Και γι' αυτό έχουμε δημιουργήσει αυτή την ομάδα εμπειρογνωμόνων AI, δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης, και συμβουλευόμαστε όλους οι εμπειρογνωμόνες από τα ακαδημαϊκά Ινστιτούτα, από ε, ενώσεις χρηστών, από ενώσεις πολιτών, ώστε να φτάσουμε σε έναν ε, οδηγό, αν θέλετε, ηθικών συστάσεων και ώστε να έχουμε και κάποιες συστάσεις χρήσιμες για την ε, πολιτική ηγεσία. Η ομάδα αυτή υψηλού επίπεδου εμπειρογνωμόνων χρησιμοποιεί και ένα, μια πλατφόρμα με πάνω των 1.700 εγγεγραμμένων μελών και σας ε, καλώ να λάβετε και εσείς μέρος αυτή τη συζήτηση. Αυτή λοιπόν η ομάδα εμπειρογνωμόνων ε, συναντήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου και δημοσίευσε μία έκθεση Διακόπτεται το μικρόφωνο της ομιλήτριας εδώ. Συγγνώμη, λέει η ομιλήτρια. Ναι, επαναλάβω λοιπόν ότι η ομάδα αυτή εμπειρογνωμόνων ασχολείται με τα θέματα διαφάνειας, ευθύνης, χρήσης της τεχνολογίας αυτής. Στην έκθεση μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά τα στοιχεία. Και χειρίζονται το θέμα κατά οριζόντιο τρόπο, λέει η ομιλήτρια. Και ως προς την πολιτική και ως προς τις επενδύσεις το τμήμα δηλαδή τη δουλειά που αφορά στι επενδύσει για την οποιαδήποτε κατάχρηση τη τεχνολογία αυτή σε όλα τα χρηματοδοτούμενα προγράμματά μας υποστηρίζουμε την έρευνα και την ανάπτυξη ώστε να καλύπτουμε τα θέματα διαφάνειας. Πράγματι εδώ χρειαζόμαστε περισσότερη δουλειά προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι ασφαλές και αξιόπιστο Θα πρέπει όμως να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα επίπεδα χρηστών του συστήματος και αλλά και σχεδιαστών του συστήματος ε, θα συμμετέχουν σε μια σε δομή, σε ένα σχεδιασμό και λειτουργικού αλλά και ηθικού συστήματος. Αυτά είναι τα στοιχεία της συζήτησης προκύπτουν από την ομάδα των εμπειρογνωμόνων. Για τις καταχρήσεις αυτές ε, ή τις οποιασδήποτε κακές προθέσεις, πρέπει να πούμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την ίδια την τεχνολογία ώστε να εντοπίζει τέτοιες παρεκκλήσεις. Από μόνη της. Ήδη χρησιμοποιούνται κάποια στοιχεία της τεχνολογίας αυτής για την ε, κατάχρηση, για παράδειγμα, για τα κρούσματα στη ε, χρησιμοποίηση των τραπεζικών καρτών. Εκτός λοιπόν από τα θέματα προστασίας δεδομένων, χρειαζόμαστε μια πιο ανθρώπινη προσέγγιση στα θέματα της χρήσης τεχνολογίας αυτής. Πρέπει δηλαδή να σεβόμαστε την ιδιωτικότητα. Πράγματι είναι στον πυρήνα της προσέγγισης για τα στοιχεία δικαίου και διαφάνειας. Επίσης είναι μέρος της εντολής της ομάδας αυτής εμπειρογνωμόνων Γνωρίζουμε επίσης τα προβλήματα της εμπιστοσύνης κοινή γνώμης, είναι ουσιαστική σημασία να αναπτύσσεται. Αναφέρθηκα πριν, λέει ο Μιλήτρια, στην σημασία, συμμαχία AI. Προσπαθούμε να καταφέρουμε το κοινό να καταλαβαίνει ποια στοιχεία, ποιες συνιστώσεις του συστήματος αυτού είναι τις τεχνολογίες αυτής είναι, είναι χρήσιμες για την δραστηριότητά τους και για την ποιότητα των δεδομένων επίσης σε όλα μας τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα υποστηρίζουμε την ανάπτυξη τραπεζών δεδομένων που να είναι ασφαλείς, καθαρές και να προάγουμε την ε, ανταλλαγή των δεδομένων αυτών από τις επιχειρήσεις. Συμπερασματικά λοιπόν θα έλεγα ότι η ηθική στην τεχνική νοημοσύνη, η εθνική προσέγγιση δηλαδή, είναι ένα πλεονέκτημα, ένα προβάδισμα που έχει η Ευρώπη, όπως και στο σύστημα προστασίας δεδομένων που έχουμε. Θα πρέπει λοιπόν από κοινού και με τους χρήστες και με τους νομοθέτες να αναπτύξουμε ένα ασφαλές πλαίσιο για τη χρήση τεχνολογίας αυτής, διατηρώντας καλή ισορροπία μεταξύ της νομοθεσίας και της ωφέλειας που θα έχει αυτή η ε, τεχνολογία για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους πολίτες. Δηλαδή να μην υπερβάλλουμε ρυθμιστικώς. Ευχαριστώ πολύ. Εκεί συμμετέχουν και οι οι αξιωματούχοι προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι DPA, συμμετέχουν με κυβερνητικέ οργανώσει σε αυτή την ομάδα υψηλού επίπεδου. Ο κύριο Μπόνι κατά πάσα πιθανότητα θα γνωρίζει. Απλά ρωτάω για να το γνωρίζουν και οι υπόλοιποι. Δεν χρειάζεται να μα απαντήσετε επί μακρόν. Ένα απλό ναι ή όχι. Κομισιόν. Δεν ξέρουμε αν έχουμε αρχέ προστασία προσωπικών δεδομένων που να συμμετέχουν, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι ειδικοί επί του θέματος της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Υπάρχουν και εκπρόσωποι οργανώσεων προστασίας των καταναλωτών. Πρόεδρος, ναι, όλοι γνωρίζουν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και επίσημες αρχές που να συμμετέχουν στην ομάδα υψηλού επίπεδου. Κύριε Μπόνι, υπό το άρθρο 54 ε, η συμβολή μας ε, στην Ήτρε είναι πολύ σημαντική, βεβαίως. 8 ε, Νοεμβρίου είναι η προθεσμία. Κύριε Μπόνι, τα γνωρίζετε. Πείτε μας κι εσείς. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω πολύ για τις ε, απόψεις σας, συνάδελφοι. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι συμφωνούμε στα βασικά. Είναι πολύ σημαντικό να καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση, διότι για να μιλήσω ανοιχτά, βρισκόμαστε στο τέλος της θητείας. Δεν είναι νομοθετικού περιεχομένου το χαρτοφυλάκιο αυτό, αλλά είναι μια έκθεση για την τεχνητή νοημοσύνη που χωρίς τη δική μας συμβολή, όπως και να έχει, θα πλαισιώσει τη μελλοντική συζήτηση που θα γίνει μετά τις εκλογές. Πολιτικά λοιπόν είναι πολύ σημαντική η έκθεση αυτή. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε αυτόν τον κατακαιρματισμό. Και ο τομέας που σχετίζεται με την ασφάλεια, την προστασία της ιδιωτικότητας, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά και τα ηθικά ζητήματα, είναι ε, θέματα που μας απασχολούν ε, σε διάφορους τομείς πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν είναι φυσικά εύκολο να ξεκινήσει μια συζήτηση για αυτά τα δεοντολογικά ηθικά ζητήματα. Εγώ έχω συμμετάσχει σε συζητήσεις με εμπειρογνώμονες, με επιστήμονες, με ερευνητές και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου σαφή. Ούτε υπάρχει ομοφωνία γύρω από αυτά τα θέματα. Στα πολιτιστικά ζητήματα για παράδειγμα ή για να μην περιπλέξω περαιτέρω τη συζήτηση, απλώς να αναφέρω θρησκευτικά θέματα υπάρχουν κάποιες διαφορές από χώρα σε χώρα και γι' αυτό πρέπει να γίνει μια ανοιχτή συζήτηση και ε, καθήκον μας εδώ ως Επιτροπή ΛΥΜΠΕ είναι να θέσουμε, να αναδείξουμε τα δεοντολογικά ηθικά ζητήματα, να τα προβάλλουμε περισσότερο, να ενισχύσουμε την ευαισθητοποίηση όλων των εταίρων. Πρόσφατα η ΕΠΑ, αν, αν θυμάμαι σωστά, πριν από δύο χρόνια, αποφάσισαν στα πολυτεχνία τους να υπάρχουν τμήματα, σε, όλα τα πολυτεχνικά τμήματα, να διδάσκονται και ηθικά ζητήματα, δεοντολογικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι χρήσιμο αυτό για να δώσουμε και στην ε, Ήτρε κάποια απτά παραδείγματα για το πώς μπορούν να λυθούν ε, ή εν πάση περιπτώσει πώς μπορούμε να χειριστούμε αυτά τα ηθικά ζητήματα. Όπως και να έχει, ευχαριστώ και την Κομισιόν για την παρουσία της εδώ, για τους, τους συναδέλφους για την ε, συζήτηση, για τη συμβολή τους. Είναι πραγματικά πολύ συναρπαστική η συζήτηση αυτή. Ναι, δεν είναι περιθωριακά αυτά τα θέματα, ε, λέει ο Πρόεδρος. Ε, ούτε δευτερεύουσα σημασία θέματα. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα και που ε, άπτονται ε, άμεσα του θέματος που επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή η Επιτροπή Ήτρε. Λοιπόν, προθεσμία για τροπολογίες 8 Νοεμβρίου. Και συνάδελφοι, περνάμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε την παρουσίαση της κυρίας Κέγγε του σχεδίου Έκθεση για το θέμα τη δημιουργία ενό ευρωπαϊκού δικτύου αξιωματούχων ε, συνδέσμων για τη μετανάστευση. Ε, είστε έτοιμοι συνάδελφοι. Σεσίλ, ωραία. Σου δίνω το λόγο για να παρουσιάσει την έκθεσή σου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Κλόντο. Ευχαριστώ και την Κομισιόν για την πρόταση τροποποίησης του κανονισμού Το χρόνο που μου διαθέτετε θα τον χρησιμοποιήσω για να σας παρουσιάσω τις βασικές αλλαγές που έχω κάνει στο κείμενο. Η αξιωματική σύνδεσμη μετανάστευσης όπως έχουμε δει δεν είναι μια νέα ιδέα. Ε, από το 2004 πρωτοεμφανίστηκε και έγιναν αλλαγές το 2011 ώστε να συμπεριληφθεί και ο ευρωπαϊκός αυτός αξιωματικός και ο σχετικός οργανισμός. Έτσι ενισχύεται ο συντονισμός των αξιωματικών συνδεσμών μετανάστευσης ώστε να μπορούν πιο αποτελεσματικά να υλοποιούν τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης. Με σκοπό την έχουμε τέτοιου αξιωματικού που λειτουργούν ε, κάπως πιο τυποποιημένα. Γι' αυτό δημιουργήσαμε αυτό τον αξιωματικό σύνδεσμο που θα λειτουργεί το ίδιο ως απεσταλμένος των κρατών μελών και ως ε, ε απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θα είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι θα ασχολούνται με θέματα μεταναστευτικά και εδώ αντικατέστησα τον κατάλογο που δεν είναι εξαντλητικός όπως τον προτείνει η Κομισιόν με μια ορολογία πιο ευρεία που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του μεταναστευτικού φαινομένου. Όσον αφορά τα καθήκοντα των αξιωματικών συνδέσμων, θεώρησα ότι έπρεπε να παρουσιάζουμε περισσότερες λεπτομέρειες από όσα προτείνει η Κομισιόν, κυρίως όσον αφορά τις επαφές με τις τρίτες χώρες, όπου προσέθεσα τις τοπικές αρχές και τις αρχές της κοινωνίας των πολιτών και τους οργανισμούς κοινωνίας πολιτών. Επίσης, ε, η δράση συλλογή ε, και επεξεργασία των πληροφοριών. Επίση, οι αξιωματικοί συνδεσμοί θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουν και επιχειρησιακέ ε, δυνατότητε, γνώσει και επαφέ στι τρίτε χώρε. Πολύ μεγάλη σημασία και χρησιμότητα ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία με τι εν αλλά και για να πληρούνται κάποιε απαιτήσει πληροφοριών και διαμόρφωση ε, μεταναστευτικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταξύ των τροποποιήσεων των τροπολογιών ε, που έχω υποβάλει, αναφέρομαι στην τυπολογία των πληροφοριών που θα παρέχονται, ειδικότερα όσον αφορά το, προφίλ, το ηλικιακό προφίλ. Ε, εκεί αναφέρω τις διάφορες τυπολογίες που έχουμε διεθνώς που υιοθετούν οι τρίτες χώρες καθώς και την τήρηση γενικότερα των θεμελιωδών δικαιωμάτων Εκεί στη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων έχω επικεντρωθεί κυρίω. Παρουσιάζοντα πρώτα απ' όλα μια οριζόντια τροπολογία που αναφέρει ρητά ότι οι λειτουργίες των εξωματικών συνδεσμών θα ασκούνται με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων και ειδικότερα των πιο ευάλωτων ατόμων. εφόσον δεν έχουν επαρκή προσόντα, τα αξιωματικοί σύνδεσμοι που διορίζουν τα κρατη θα πρέπει να ακολουθούν μια κατάρτιση επαρκή για την αντιμετώπιση των ε, ευαίσθητων ανθρώπων, ειδικότερα των γυναικών, των ευάλωτων ε, κατηγοριών, κυρίως των γυναικών και των ανηλίκων. Θα πρέπει να είναι ειδικοί στην, σε θέματα προστασίας των ε, ανηλίκων και ίσης μεταχείρισης των φύλων. Στο steering board έχω προσθέσει τη δυνατότητα το κοινοβούλιο επιδαλώντας το ρόλο του ως συνομοθέτη θα πρέπει να μπορεί να καλείται ως παρατηρητής στις σχετικές συνεδριάσεις. Ελπίζω λοιπόν ότι η Επιτροπή και τα κρατημέλη δεν θα φέρουν αντίρρηση γι' αυτό. Έτσι έχω προβλέψει το Κοινοβούλιο να λαμβάνει ε, τις προτεραιότητες και τις δραστηριότητες ε, που περιλαμβάνονται στο διαιτές πρόγραμμα. Μιλάμε για σημαντικές πηγές πληροφοριών όσον αφορά τις δραστηριότητες του δικτύου. Εδώ στο Κοινοβούλιο, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτά. Ε, εμπιστεύω, αναθέτω λοιπόν, έχω εμπιστοσύνη στους σκιώδεις συζητητές και είμαι και ανοιχτή για συζήτηση με το Συμβούλιο και την Κομισιόν, ώστε το συντομότερο δυνατόν να υιοθετήσουμε αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε, Σεσίλ. Πάμε στους Κιώδης για το ΕΛΚΑ. Αλεσάνδρα Μουσουλίνη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ, όπως είχα και την ευκαιρία να πω ε, στην αρχή, βρίσκω θετικό το να δημιουργήσουμε μια, έναν τέτοιο πιο ευρωπαϊκό θεσμό, έναν τέτοιο αξιωματικό η εισηγήτρια διαγράφει τις σχετικές ε, παραγράφους ε, που αναφέρονται στα κράτη-μέλη, τους οργανισμούς ε, και τα θεσμικά όργανα. Τώρα, απέναντι στις οργανώσεις των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών που ενισχύουν την διασύνδεση με το ήλος, το σημείο που κατά την άποψή μου ίσως να ενέχει έναν κίνδυνο είναι ότι στο σχέδιο της εισηγήτριας τελικώς αυτός ο θεσμός, αυτός ο αξιωματικός αποδυναμώνεται γιατί είναι προφανές ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι εξαιρετικά σημαντικά και ήδη η Κομισιόν αναφέρεται στην υποχρέωση συμμόρφωσης προς τα θεμελιώδη αυτά δικαιώματα αλλά η διαρκής αναφορά και η διαγραφή των στόχων των αντικειμένων ύλος που είναι για τη μετανάστευση, τον επαναματρισμό και τη διευκόλυνση όλων αυτών των διαδικασιών καθίστανται κάτι διαφορετικό, κάτι πιο αφηρημένο. Σαν επιτηρητές των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων. και εκεί έχουμε αλληλεπικαλύψεις ή και συγκρούσεις με την εντολή της ε, ΕΑΣΟ. Οι αξιωματικοί αυτοί ορίζονται από τα κράτη-μέλη, την Κομισιόν και τους οργανισμούς. Εάν εμείς αποδυναμώσουμε, τροποποιήσουμε τέλος πάντων την εντολή τους, τους βάλουμε να κάνουν κάτι άλλο, τότε δεν ε, συμμορφούμαστε και προς την ε, επικουρικότητα ως προς το κράτος μέλος. Δηλαδή αναθέτω με διαφορετικές εντολές σε διαφορετικά πρόσωπα. Επίσης αυτή η διαρκής αναφορά στα θεμελιώδη δικαιώματα σημαίνει ότι εκεί που δεν το κάνουμε είναι σαν να μην τα παρακολουθούμε. Εάν λοιπόν από την αρχή θα μπορούσαμε να έχουμε μια τοποθέτηση στήριξης σε μια εντολή λίγο πιο ευρωπαϊκής φύσεως δεν θα, θα αποκλίνουμε λιγάκι από, το, από τη βασική κατεύθυνση στόχευση των ε, αξιωματικών αυτών. Σας ευχαριστώ λέω Για τους άλλους σκιώδεις, Άλντε και Πράσινη δεν είναι εδώ. Γκούε, Μαρή Κριστίν Βεργιά, παρακαλώ ή μήπως θέλετε να τοποθετηθείτε και εκ μέρους Άλντε, η Σοφή θα μας μιλήσει εκ μέρους ε, της Άλντε, παρακαλώ. Ναι, πρόεδρε, η κυρία Γκρισμπέκ μου ζήτησε να διαβάσω τη δήλωσή τους που λέει θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την απουσία μου και να ευχαριστήσω την ε, Σοφή, εμένα, την ίδια δηλαδή, για τη διαβίβαση αυτού του μηνύματος. Ευχαριστώ την Σεσίλ για τη δουλειά και για την ε, πρόταση κομισιών. Πολλοί μας ικανοποιούν οι υποβολές τροπολογίας της κυρίας Κιέγκε για πρόσθετα εχέγγυα προς τα θεμελιώδη δικαιώματα για το δίκτυο αυτών των ILO. Ιδιαίτερα σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών, ε, πολύ μας ικανοποιούν οι σχετικές αναφορές, όπως και η δυνατότητα του, της, ε, που δίνεται μέσα από το κείμενο της τροπολογίας 29. Αυτοί οι ILO θα πρέπει να έχουν έναν ενεργή ρόλο στο πλαίσιο του μεταναστευτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και απέναντι στις τρίτες χώρες, υπό την έννοια αυτή, η τροπολογία 24 μας φαίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Θα ήθελα να ζητήσω όμως μάλλον να διαβαστεί το μήνυμα προς τον Κομισιόν, όπως είχαμε συζητήσει στην προηγούμενη συνέντευξη σκιωδών, χρειαζόμαστε πρόσθετα εχέγγυα και μηχανισμούς στήριξης, ώστε να είναι το κείμενο επαρκώς σαφές σχετικά με τη διασύνδεση μεταξύ των κρατών μελών και των ILO. Δεν θα πρέπει δηλαδή όλα αυτά να είναι απλώς ένα κενό γράμμα αποκρύπτοντας τα κρατημέλη ενδεχομένε πληροφορίες από τους αξιωματικούς αυτούς για να διατηρήσουν, να διαφυλάξουν αν θέλετε τα συμφέροντά τους. Ευχαριστώ πάντως ε, για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε και μάλιστα σε πολύ στενά χρονικά περιθώρια. Σας ευχαριστώ Σοφή. Η Μαρή Κριστίν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τη συνάδελφο τη ΕΣΥΛ. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με όλες τις προτάσεις και τις τροπολογίες. Το θέμα αυτό, καθώς και η διαδικασία που έχει ξεκινήσει η Κομισιόν, αν κατάλαβα καλά, θα μας βοηθήσει να έχουμε μια ολιστική αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος. Πιστεύω ότι είναι καλή η προσέγγιση αυτή. Από το 2015 και 2016 ε, βγαίνουμε έχοντας καταφέρει να βάλουμε κάποια λογική στις μεταναστευτικές μας πολιτικές. Αλλά λέγοντας αυτό δεν θέλω να ε, συζητάμε μόνο τις ε, εντός εισαγωγικών προβληματικές ε, χώρες στο νότο της Μεσογείου. Την περασμένη εβδομάδα λάβαμε τα επίσημα νούμερα για τις άδειες ε, παραμονής που έχουν εκδώσει τα κράτη-μέλη για μακροχρόνιες διαμονές και για τρίτη συνεχή χρόνια. Οι Ουκρανοί είναι η πρώτη που, σε αριθμό που λαμβάνουν τέτοιες άδειες παραμονής. 500.000 πέρυσι, 662 φέτος. Είναι η μεγαλύτερη μεταναστευτική ροή που έχουμε, δεν είναι σε σχέση με το θέμα αυτό. Καμία άλλη χώρα δεν έχει στείλει τόσους πολλούς μετανάστες. Ε, ε, και ε, σε μεταναστευτική κίνηση τώρα. Προτιμώ τη λέξη κίνηση από τη λέξη ροή. Εγώ λοιπόν θα προτείνω κάποιες τροπολογίες που να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη αυτή την ισορροπία. Όχι λοιπόν να έχουμε μια έμονη ιδέα μόνιμα παρότι είναι σημαντικές τις μεταναστευτικές κινήσεις από τον νότο που ονομάζονται και παράτυπες. Ε, με τη Σεσίλ συμφωνούμε ε, στο ότι αφού μιλάμε για παράτυπες μεταναστεύσεις εδώ, παράτυπες κινήσεις, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουμε νόμιμες οδούς μετανάστευσης, οπότε θα πρέπει να κάνουμε και μια σύγκριση μεταξύ των χωρών που δεν διαθέτουν τακτικές οδούς μετανάστευσης και των χωρών που διαθέτουν. Και δεν έχω τίποτα κατά των Ουκρανών. Χαίρομαι που ένα σωρό Ουκρανοί έρχονται εδώ να δουλέψουν ε, στην Πολωνία γιατί το 87% αυτών των αδειών παραμονή ε, είναι άδειε εργασία. Οπότε μιλάμε για οικονομικού μετανάστε ε, και το 85% αυτών των Ουκρανών έρχονται να δουλέψουν στην Πολωνία. Οπότε χαίρομαι. Αλλά θέλω και αυτό το ζήτημα να το συζητήσουμε. Και συζητώντα και του αξιωματικού συνδέσμου να έχουμε μία ε, ολική εικόνα του μεταναστευτικού ζητήματος. Επίσης κάτι άλλο που θέλω να, στο οποίο θέλω να επιμείνω, να κοιτάμε τις αφήξεις αλλά και τις αναχωρήσεις. Αλλά αν έχουμε 1,5 εκατομμύριο ε, Ουκρανού που φτάνουν στην Πολωνία, γιατί σήμερα νομίζω 1,5 εκατομμύριο είναι οι Ουκρανοί που ζουν στην Πολωνία. Είμαι πεπισμένη παρόλα αυτά ότι και κάποιοι φεύγουν. Αυτά τα ρεύματα αποχώρηση δεν τα εξετάζουμε όπως δεν εξετάζουμε και τους Ευρωπαίους που μεταναστεύουν σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε χρειαζόμαστε μια τέτοια συνολική εικόνα. Αυτή η εξωματική σύνδεσμοι λοιπόν πιστεύω θα μπορέσουν να μας χρησιμεύσουν στα θέματα αυτά. Τέλος, ε, είχα μια ερώτηση σε σχέση με τις τροπολογίες της ΕΣΥΛ. Πρόσθεσε το ζήτημα των, των προγραμμάτων μελλοντικών ε, μετακινήσεων. Θέλω να μου πει τι σημαίνει να καταλάβω καλύτερα. Επίσης άλλο ένα θέμα για το οποίο θα υποβάλω τροπολογίες είναι η προστασία των δεδομένων. Θα, τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να προστατεύονται αλλά να έχουμε και ανανυμοποίηση των ε, στοιχείων, των ονομαστικών στοιχείων που μας βοηθούν να καταλάβουμε τις μεταναστευτικές ροές. Τέλος, όσον αφορά την ενίσχυση του διαλόγου με τις τρίτες χώρες, πιστεύω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε στο ότι κάποιε τρίτε χώρε ε, σέβονται και τηρούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικότερα, άλλε όχι. Αυτό το ζήτημα λοιπόν τη συνεργασία και του διαλόγου, ε, τη ενισχυμένη συνεργασία και του ενισχυμένου διαλόγου θα πρέπει να λαμβάνει και αυτή την παράμετρο υπόψη κάποιε χώρε. Πιστεύω είναι χώρε ε, με τι οποίε ενισχύουμε το διάλογο και τη συνεργασία για τη μετανάστευση για να κατανοήσουμε τι βαθιέ ε, αιτίε της μετανάστευσης ε, και εκεί συναντάμε κάποια προβλήματα ε, που θα πρέπει να μας απασχολήσουν να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτές τις χώρες το οποίο οδηγεί στη δημιουργία αυτών των ροών. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Μήπως σε λίγη Κομισιόν να προσθέσει κάτι. Πολύ σύντομα σας παρακαλώ όμως. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, άκουγα την γαλλική διερμηνία και υπήρχε μια μικρή καθυστέρηση. Ένα ερώτημα δέθηκε προς την Κομισιόν σχετικά με το πώς θα εξασφαλιστεί η υποχρέωση διαμοιρασμού πληροφοριών που βρίσκονται στην πλατφόρμα, όπως εμφανίζεται στο κείμενο. Και όπως έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, πιστεύουμε ότι το άρθρο 5 με το να χρησιμοποιεί αυτό τον όρο «σαλ» ε, αποτελεί επαρκές εχέγγυο. Δεν έχουμε όμως αντίρρηση να ενισχύσουμε αυτήν την ενθάρρυνση των κρατών μελών για τον διαμοιρασμό από πλευράς κρατών μελών των πληροφοριών και την ε, διάθεση των πληροφοριών αυτών στην πλατφόρμα. Ευχαριστώ. Σεσίλ, να κάνεις τις καταληκτικές παρατηρήσεις, σε παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ όλους ε, για την ε, συνεισφορά τους. Είμαι σίγουρη ότι θα ξανασυναντηθούμε, θα ξανασυζητήσουμε και τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί και τις διαφορές που ενδεχομένως να υπάρχουν. Και επιχειρώ να απαντήσω ήδη σε ένα σημείο αυτό που αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά που τοποθετήσαμε στο κείμενο δεν αποδυναμώνουν ούτε τροποποιούν τα καθήκοντα και την εντολή του αξιωματικού. Αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά την άποψή μου δεν μπορούν να αποσπώνται από το μεταναστευτικό φαινόμενο. Επιχειρήσαμε να επανασυνδέσουμε λοιπόν την πτυχή αυτή γιατί τη θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική. Στο κείμενο τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρονται απλώς ή στα πλαίσια αιτιολογικής σκέψης. Επιχειρώντας ακριβώς να επαναφέρουν το θέμα αυτό. Όμως διατηρείται απολύτως η λειτουργία και η εντολή του ILO. Για την ΕΑΣΟ θα είναι μεταξύ άλλων και καθήκον της Κομισιόν να διευκρινίζει τις ε, σχετικές αρμοδιότητες, διότι μέχρι σήμερα οι υπάλληλοι Τη ΕΑΣΟ είναι ελάχιστη και δεν θα μπορούσαν να καλύψουν το σύνολο της επικράτειας. Και θα έκλεινα και, απευθύνοντας και μια ερώτηση και πολύ με ικανοποιεί ε, και η αναφορά της ε, Άλντε στους ανήλικους γιατί ακριβώς ήταν και δική μας πρόθεση να ενισχύσουμε την προστασία των ευάλωτων ομάδων μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά. Η Μαρία Κριστίνα αναφέρθηκε σε θέματα κινητικότητας. Εγώ ανέπτυξα τροπολογίες σημειώνοντας ότι υπάρχουν ότι και στο Αγκαντές φτάνουν άτομα, άνθρωποι που μένουν εκεί μπλοκαρισμένοι. Δηλαδή θα πρέπει να δει κανείς πού μπορούν να πάνε αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να περιοριστούμε στην Ευρώπη ή να δούμε το θέμα ευρύτερα με πιθανές, πιθανούς προορισμούς που θα μπορούσαν να έχουν οι άνθρωποι αυτοί που αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες αυτές. Δηλαδή όλα αυτά θα ήταν ενδιαφέρον να τα γνωρίζουν και όλοι αυτοί που μετακινούνται. ώστε να μην μένουν εκρεμή και μπλοκαρισμένα τα άτομα, αν θέλετε, μεταξύ ε, διαφορετικών εδαφών. Ευχαριστούμε Σεσίλ για τη δουλειά σου. Ευχαριστώ και τους Σκιώδης. Καλή επιτυχία με τις μελλοντικέ συνεδριάσεις σας. Προθεσμία τροπολογίες είναι ε, η 19η Νοεμβρίου. Σας ευχαριστώ όλους για τη δουλειά σας, συνάδελφοι. Και πάμε στο επόμενο θέμα. παρουσίαση σχεδίου έκθεσης για την μεταρρύθμιση του συστήματος πληροφοριών θεωρήσεων. Κάρλος, είσαι έτοιμος? Ωραία. Δίνω λοιπόν το λόγο αμέσως στον κύριο Κουέλιο για να μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσής του. Κάρλος, παρακαλώ. Ευχαριστώ, θα μιλήσω πορτογαλικά. Ευχαριστώ λοιπόν Επαναλαμβάνω ότι το Σέγγεν και η ελευθερία κυκλοφορίας αποτελούν τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. και συνοδεύονται βεβαίως από μέτρα που εγγυώνται την ασφάλεια στα κοινά μας σύνορα και την συνεργασία των αστυνομικών ε, δυνάμεων στην επικράτεια των κρατών μελών μας. Η Σέγγεν και η ελευθερία κινήσεων απαιτούν κοινή πολιτική θεωρήσεων που θα εξασφαλίζουν τις ελευθερίες αλλά και την ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίζεται δηλαδή ότι οποιοδήποτε διέρχεται από τα σύνορά μας, είτε για επίσκεψη, είτε για σπουδές, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, θα δεσμεύεται από αυτά τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο VIS. Μιλούμε δηλαδή για την χορήγηση θεωρήσεων που θα ε, εμποδίζει το visa shopping από ε, προξενικές αρχές, συνοριοφύλακες σε όλη την Ευρώπη. Διότι αυτό το φαινόμενο το παρατηρούμε σε όλα τα προξενία των κρατών μελών και στα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σέγγεν. Μιλάμε μόνο για θεωρήσεις ε, μικρής διάρκειας για τουριστικούς σκοπούς. Το 2017 60, 60 εκατομμύρια τέτοιες θεωρήσεις χορηγήθηκαν. Ωστόσο, στον Σέγγεν δεν εισέρχονται μόνο ε, τουρίστες, αλλά και φοιτητές, ε, ερευνητές, εργαζόμενοι ή και συγγενείς ανθρώπων που έχουν δικούς τους εδώ στην Ευρώπη. Όλοι αυτοί λοιπόν καταγράφονται στο σύστημα VIS. Σύμφωνα με τη Eurostat, πέρσι ένα εκατομμύριο άτομα μετανάστευσαν προς την Ευρώπη για να εργαστούν. Και πάνω από 800 ε, ε, ήρθαν για επίσκεψη. Πάνω από ένα εκατομμύριο ήρθαν για να φοιτήσουν. όλοι αυτοί δεν καταγράφονται πουθενά σε καμία βάση δεδομένων. Είναι μια κατάσταση στην οποία και εγώ αλλά και η Άννα έχουμε ασκήσει κριτική. Υπάρχει και αυτό το φαινόμενο της χρυσή βίζας που επίσης τα στοιχεία αυτών που, που λαμβάνουν αυτές τις θεωρήσεις δεν καταγράφονται στο VIS ούτε υπάρχει απόλυτη συμβατότητα μεταξύ των πληροφοριών Σέγγεν και των πληροφοριών θεωρήσεων. Και αυτά όλα θέλουμε να αλλάξουν. Αν θέλει κάποιο Καναδό να μεταναστεύσει στην Ευρώπη, τότε δεν μας ενδιαφέρει πού θα εγκατασταθεί η θεώρησή του θα πρέπει να καταγράφεται στο VIS. Είτε πάει να μείνει στην, ε, στο Βέλγιο, είτε πάει να μείνει σε κάποια άλλη ε, ευρωπαϊκή χώρα. Θα πρέπει τα δεδομένα αυτά να είναι ανακτήσιμα πάντοτε. Μα με αυτόν τον τρόπο άλλωστε εξασφαλίζεται και η ελεύθερη κυκλοφορία του. Αλλά πλέον ξεκαθαρίζεται ότι η θεώρηση έχει και μια πολύ σημαντική διάσταση ασφάλειας. Αυτή η διάσταση μάλιστα στο μέλλον θα ενισχύεται όλο ένα και περισσότερο. Ενδέχεται να υπάρχουν άνθρωποι που θα θέλουν να εγκατασταθούν ε, να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ευρώπη. Για να μην χρειάζεται λοιπόν κάθε φορά να περνάνε, διαρκώς να περνάνε από ελέγχους αυτοί οι άνθρωποι, είναι πολύ σημαντικό οι πληροφορίε που συνδύονται με τη θεώρησή του να είναι καταγεγραμμένες και αυτόματα να μπορούν, να μπορούν οι αρχέ να τι ανακτούν και να έχουν πρόσβαση σε αυτέ. Βεβαίω πάντοτε λαμβανομένων υπόψη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όμω πρέπει στα νομικά μα κείμενα να ξεκαθαρίζουμε ότι θα υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει και χειροκίνητο έλεγχο ανα πάσα στιγμή. Πάλι βεβαίως με προστασία της ιδιωτικότητας των ατόμων, πάντοτε. Υπάρχουν και οι αρμόδιες υπηρεσίες άλλωστε και προβλέπονται, που πρέπει να, να δημιουργηθούν, να ιδρυθούν στα κράτη-μέλη. Βεβαίως, επίσης, θα πρέπει να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι πριν από τη χορήγηση της θεώρησης. Δεν είναι λογικό αυτό που προτείνει η Κομισιόν. Άνθρωποι να υπάγονται σε αυτούς τους ελέγχους αφού τους δοθεί η θεώρηση οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να γίνονται εκ των προτέρων. Έχουμε πει επανειλημμένως ότι αυτές οι αρχές θα πρέπει να διαπνέουν και το VIS και το SIS και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε ε, την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού του Σέγγεν και της ελεύθερης κυκλοφορίας. Είναι σημαντικό επίσης το VIS να μπορεί να προσαρμόζεται σε τυχόν αλλαγές των καταστάσεων, σε εξελίξεις που θα υπάρχουν. Υπάρχουν τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες διαδικτυακές επιθέσεις που πολύ συχνά συνδέονται και με πολιτικούς κινδύνους που άπτονται του θέματος της κεντρικής αποθήκευσης όλων αυτών των δεδομένων. Όλα αυτά μέχρι στιγμής ήταν ε, ε, υποχρέωση των κρατών μελών. Τα ίδια ισχύουν και για τον Ιουλίζα, τον οργανισμό που είναι αρμόδιος για την προστασία των δεδομένων. Χρειαζόμαστε χρονοδιάγραμμα, συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασιών και δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έχει ε, προταθεί από την Κομισιόν, ούτε καν η δυνατότητα ε, υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων. Νομίζω ότι αυτό είναι, δεν, είναι, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Πρέπει να ενισχυθούν οι μηχανισμοί ελέγχου του Κοινοβουλίου και η λογοδοσία βεβαίως, υποχρέωση λογοδοσίας της Κομισιόν. Εγώ προτείνω να οριστεί η προθεσμία διετής για την υλοποίηση όλων αυτών, αντί της λευκής επιταγής που μας ζητάει η Κομισιόν. Συνάδελφοι, Σα ευχαριστώ λοιπόν που είχα την ευκαιρία να σα παρουσιάσω αυτό το σχέδιο έκθεση. Είμαι βέβαιο ότι σε συνεργασία με του Σκιώδης θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τη θέση του Κοινοβουλίου. Βεβαίω είναι περίπλοκη η έκθεσή μα αυτή, Όμω το γνωρίζουμε επίση ότι βρισκόμαστε στο τέλο τη ε, κοινοβουλευτική θητεία και από αυτή την άποψη βεβαίω πρέπει γρήγορα να ολοκληρώσουμε τι διαπραγματεύσει. Έχουμε ήδη κάνει κάποιε τεχνικέ συνεδριάσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στι 20 Νοεμβρίου θα ε, γίνει η πρώτη συνεδρίαση των σκηνοδών ε, εισηγητών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε Κάρλος και ευχαριστούμε και για την πολλή δουλειά σε αυτόν τον ε, πολύ σημαντικό φάκελο. Για τους κοιόδης τώρα. Η Birgit θα εκπροσωπήσει τον τον κύριο Νίντα Μιούλε που είναι ο Σκιώδης. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την Κομισιόν για την ε, πρόταση και τον κύριο Κοέλιο για το σχέδιο. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό σημείο εκκίνησης για τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν. Καθότι ο κύριος ε, Νίντα Μιούλε δεν μπορούσε να είναι μαζί μας εδώ σήμερα, θα αναφερθώ σε κάποιες από τις πτυχές που επισημαίνει. Έχουμε ακόμα κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα να συμπεριληφθούν τα δεδομένα των μακροπρόθεσμα διαμενόντων στο σύστημα θεωρήσεων. Επίσης έχουμε ανησυχίες για την μείωση της ηλικία για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμένων για τα παιδιά και τα δικαιώματα ε, σε αντιστάθμιση ιδιαίτερα στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας. Εξετάζουμε προτάσεις τροπολογίας να, που θα, επιβάλλουμε, θα υποβάλλουμε με σε αυτά τα θέματα, αλλά θα συνεργαστούμε επικοδομητικά με τον εισηγητή για να βρούμε λύσεις σε, στα ζητήματα αυτά που εκκρεμούν. Ευχαριστώ. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστώ και εγώ. Η κυρία Βεωζιά, όχι. Η κυρία Γκόμης. Παρακαλώ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κουέλιο και εγώ με την σειρά μου για την δουλειά από αυτή και τις προτάσεις που απορρέουν από τη δουλειά της ομάδας μελέτης, μάλλον της ομάδας ελέγχου Σέγγεν. Γιατί και εγώ είχα τη χαρά να συμμετέχω τέχος στην ομάδα αυτή, τη οποία προείδρευσε ο κ. Σημείωσα με ενδιαφέρον ότι θα μας ε, κάνει κάποιες προτάσεις σχετικά με αυτές τις ε, ούτως αποκαλούμενες ε, χρυσές θεωρήσεις. Είναι ενδιαφέρον, αλλά είναι το ελάχιστο θα έλεγα για την ασφάλειά μας, αλλά είναι και το ελάχιστο υπό την έννοια του δικαίου, της ισότιμης μεταχείρισης το να εισάγονται αυτές τι περιπτώσεις στις ε, τράπεζες δεδομένων. Αλλά έχω την εξή απορία. Υπάρχουν αρκετές χώρες που παραλίλω προς αυτά τα συστήματα θεωρήσεων χρησιμοποιούν ακόμα ένα σύστημα επανένωση οικογενειών ακόμα λιγότερο συντονισμένο από τις, ε, αυτές τις χρυσές θεωρήσεις. Δηλαδή πέραν αυτών υπάρχουν και άλλες δυνατότητες επανένωσης και εκεί σε αυτό το πεδίο δεν ε, υπάρχει πολύ λίγη αν όχι ανύπαρκτη συνεργασία και κανείς έλεγχος και δεν ξέρω αν αυτό το αναφέρετε στην πρότασή σας. Επίσης ένα άλλο στοιχείο που εμείς πάντοτε σημειώναμε στην ομάδα ελέγχου Σέγγεν είναι ότι είναι δύσκολο να ελέγχονται η, να ελέγχεται η έκδοση εθνικών θεωρήσεων γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται στις τράπεζες δεδομένων. Ούτε ελέγχει η Κομισιόν τα στατιστικά δεδομένα. Για παράδειγμα μεταξύ Μάλτας και Λιβύης. Όταν η Μάλτα έκλεισε την πρεσβεία της στην Λιβύη δεν είχαμε πλέον από εκείνη τη στιγμή και μετά στατιστικά δεδομένα. Αλλά συνέχισε να λειτουργεί αυτό το, θέμα, το σύστημα πωλήσεως διαθέσεως εμπαστός θεωρήσεων. Δεν δηλαδή, διελάμβανε κανείς μια τέτοια θεώρηση και μετά έπαιρνε ένα σκάφος και πήγαινε σε άλλο κράτος μέλος Έγγελ. Και εκεί δεν έλεγχε κανείς. Όχι μόνο δεν έλεγε κανείς, ούτε καν τα στατιστικά δεν ελέγχαμε. Επ' αυτόν τι μπορούμε να κάνουμε. No one else the floor, so just ask Carlos, do you want Κάρλος, ε, να σας ρωτήσω αν έχετε να κάνετε κάποια σχόλια. Α, όχι, συγγνώμη. Συγγνώμη. Η Κομισιόν θέλει να προσθέσει κάτι. Ναι, ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τα μέλη. Πρέπει να πω, οι θεωρήσει είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για πολλά κράτη-μέλη όσον αφορά την υλοποίηση τη δική μα πολιτική θεωρήσεων. Περίπου 16 εκατομμύρια θεωρήσεις έγκεν εκδίδονται κάθε χρόνο ένα εκατομμύριο κινήσεις. Ε. Πρέπει να βελτιωθεί αυτό το σύστημα, αυτός είναι ο στόχος της πρότασης αυτής ε, της Κομισιόν. Μαζί με το σύστημα εισόδων-εξόδων, το ETS ε και το VIS θα ελέγχονται πιστεύουμε καλύτερα οι υπηκοίτροι των χωρών που εισέρχονται στο χώρο Σέγγεν. Όπως είπα είναι σημαντικό η εξέλιξη, η αναβάθμιση αυτού του συστήματος πληροφοριών Σέγγεν να γίνει ε, βάσει των αρχών διαλειτουργικότητας που συζητείτε εδώ στην Επιτροπή σας και στους τριμερείς διαλόγους και θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα, όλες οι συνιστώσεις της διαλειτουργικότητας. Υποστηρίζουμε επίσης και τον εισηγητή που περιλαμβάνει τις πληροφορίες για μακροχρόνιες άδειες παραμονής και θεωρήσεις. Ε, σημειώνουμε τη διαφορετική προσέγγιση για τους ελέγχους αυτών των εγγράφων. Αναμένουμε να συζητήσουμε τα ζητήματα αυτά, όπως και όλα τα υπόλοιπα που αναφέρθηκαν στους τριλόγους, ε, το συντομότερο δυνατόν. Στους τριλόγους αυτούς θα συζητήσουμε το πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με αυτή την πρόταση νομοθετικά. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε. Κάρλος, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, και για την εξαιρετική του συνεργασία στο πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Για να απαντήσω στις ερωτήσεις της Αναγκόμες, στην εκθέσή μου σαφώς υπάρχουν αλλαγές ως προς την πρόταση της Κομισιόν. Έχουν ήδη συνταχθεί ώστε να συμπεριληφθούν οι οικογένειες. Το πρώτο δηλαδή θέμα που, έθεσε η Αναγκόμες ε, περιλαμβάνεται σαφώς στη δική μου πρόταση. Επίσης, ε, τα όσα αναφέρατε για τα στατιστικά στοιχεία και τις εθνικές θεωρήσεις. Και αυτά θεωρούμε, σκοπεύουμε, συγγνώμη, να υποχρεώνουμε τα κράτη-μέλη να ελέγχουν το σύστημα για θέματα ασφαλείας ε, και για το θέμα των θεωρήσεων ασφαλείας. Εμείς εξετάζουμε τώρα τις νομικές λεπτομέρειε για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το συμπεριλάβουμε αυτό στον κανονισμό. Ελπίζω να μην χρειαστεί να έρθουμε σε αντιπαράθεση με το Συμβούλιο, διότι εξετάζοντας το πρόβλημα σε βάθος, όλοι αντιληφθήκαν ότι δεν έχει νόημα να ελέγχουμε το σύστημα αφού εκδοθεί η θεώρηση, αλλά πριν. Αυτό έχω συμπεριλάβει και εγώ στη δική μου έκθεση. Και ελπίζω να έχω την υποστήριξή σας. Ευχαριστούμε, Κάρλος. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι πόσο σημαντική είναι η δουλειά της Επιτροπής μας. Οπότε θέλω να σας ευχαριστήσω για τις σκληρές σας προσπάθειες και σας φυσικά και του σκιώδεις. Νέα προθεσμία για τις τροπολογίες η 13η Νοεμβρίου αντί για την αρχική που ήταν η 9η. Επαναλαμβάνω τι ευχαριστή μου προς τον εισηγητή και τους συναδέλφους που πήραν τον λόγο. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο σημείο 8. Είμαστε πιο νωρίς ε, σε σχέση με το πρόγραμμα. Είναι εδώ ο εισηγητής. Ε, ε, δέχεστε να προχωρήσουμε. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνουμε και ένα διάλειμμα αρκετά πριν τις ψηφοφορίες που έχουμε σήμερα το απόγευμα που φαίνεται ότι θα διαρκέσουν αρκετά. Αν το επιτρέπει λοιπόν ο εισηγητή, θα μπούμε λίγο νωρίτερα στο επόμενο σημείο τη ημερησία διάταξη, το σχέδιο γνωμοδότηση για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιδών Δικαιωμάτων. Ο εισηγητή, ο κύριο Ντε θα παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότηση του. Κύριε Ντε παρακαλώ. Uh, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι στη γνωμοδότηση αυτή δυσκολεύτηκα λίγο με τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούσα να χρησιμοποιήσω. Είναι αρκετά συνοπτική η έκθεσή μου, τόσο όσον αφορά την ουσία της, όσο και όσον αφορά το, το έργο που έχει κάνει η Επιτροπή μας. Στην ΑΦΚΟ υπήρξε ένα μεγάλο χρονοδιάγραμμα με πολλά έγγραφα εργασίας, έχει συζητηθεί επί μακρόν, τα, τα εξέτασα όλα αυτά με μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά μου ήταν ξεκάθαρο ότι τελικά το βασικό θέμα δεν είναι ο σεβασμός του χάρτη δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη, αλλά όσο ε, ο, η, ο σεβασμός των, ε, δικαιωμάτων από τα, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπάθησα λοιπόν να ακολουθήσω και να παρακολουθήσω το, τη γραμμή της σκέψης της ε, ΑΦΚΟ ε, και τους τομείς που έχει αναδείξει η Επιτροπή αυτή. Όλα αυτά ε, ε, προκύπτουν και από τα έγγραφα εργασίας που έχει υποβάλει ο συγητής, που, που ορίζουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Για παράδειγμα, πόσο προσοχή δίνεται πέραν του χάρτη, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα κοινωνικά δικαιώματα, ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας και ο Χάρτης των Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Δεύτερον, ποιος είναι ε, η σχέση του χάρτη αυτού με την κοινωνικο-οικονομική διακυβέρνηση. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό που έχει απασχολήσει την Επιτροπή ΑΦΚΟ. Και τρίτον, η εφαρμογή του χάρτη από τους ίδιους τους οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέταρτον, ποια ένδικα μέσα έχουν στα χέρια τους οι πολίτες σε ε, περιπτώσεις παραβίασης των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων από επιχειρήσεις. Και τέλος, ερεσιμότητα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Εδώ έχει γίνει πολλή συζήτηση, αλλά σημειώνω ότι είναι και αυτό ένα σημαντικό θέμα που έχει συζητηθεί στην ΑΦΧΟ και που θα πρέπει να τοποθετηθούμε και εμείς. Λοιπόν, Έχω υποβάλει αρκετέ τροπολογίε στην έκθεσή μου και παρακινώ και τους άλλους ισχυώδεις συζητητέ, να κάνουν το ίδιο γιατί υπάρχουν πραγματικά πολλά θέματα τα οποία πρέπει να καλύψουν μέσω αυτή τη γνωμοδέτησης. Για παράδειγμα, ζητήματα που πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν είναι η μελέτη επιπτώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, κάποιες φορές οι νομοθετικές προτάσεις της Κομισιόν ε, συνοδεύονται κάποιες από τέτοιε αξιολογήσει, από άλλε φορέ όχι. Πρέπει πλέον αυτό να γίνει μόνιμο. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχει μια πραγματική, ε, μια συστηματική προσέγγιση όσον αφορά τη μελέτη επιπτώσεων ε, σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Επίσης, θεωρώ ότι αυτές οι μελέτες επιπτώσεων μπορούν να υπερβαίνουν και τα σημερινά όρια. Θεωρώ ότι ο οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων καλό θα ήταν όποτε ανα, ε, αναδιατυπώνεται ή τροποποιείται ο, ο σχετικός κανονισμός που τον διέπει, να γίνεται ρητή αναφορά στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και να υπάρχει και ένας κώδικας διοντολογίας για το προσωπικό αυτού του οργανισμού σε σχέση με το πώς χειρίζονται τα ζητήματα παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων. Από αυτή την άποψη λοιπόν βρισκόμαστε στην αρχή μιας ε, ελπίζω πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που θα καταλήξει σε μια πολύ καλή γνωμοδότηση. Αυτή που σας παρουσίασα σήμερα δηλαδή. Πρόεδρος, μίλησα εισαγωγικά για την εφαρμογή του χάρτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ε, ε, στην πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλλον παρασύρθηκα, γιατί χαίρομαι πολύ με αυτά τα θέματα. Ξέρετε, μερικές φορές ε, με συναρπάζουν ακόμη και τα πλέον βαρετά θέματα. Να το ξεκαθαρίσω λοιπόν ότι μιλάμε για κάτι πολύ πιο περιορισμένο. Μιλάμε για το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει έναν θεσμικό χαρακτήρα λοιπόν ε, γι' αυτό άλλωστε είναι καθήλυνα αρμόδια επιτροπή και η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εμείς γνωμοδοτούμε. Παρ' όλα αυτά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να καταλήξετε σε μια καλή γνωμοδότηση από την πλευρά της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Ποιο θέλει το λόγο, η Ρομπέρτα. Ευχαριστώ. Ε, αντικαθιστώ την Μπάρμπαρα Ματέρα που, μας, που μου άφησε κάποιες σημειώσεις τις οποίες και θα διαβάσω. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ντε για, το, για τη δουλειά του. Η τελική έκθεση της ΑΦΚΟ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη και βασίζεται ακόμα στο έγγραφο εργασίας. Η έκθεση εφαρμογής θα αναδείξει ε, το ρόλο του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων ως πρωτογενές δικαίου όσον αφορά τους οργανισμούς και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ως ΛΥΜΠΕ ε, βεβαίως ε, είμαστε απόλυτα προσελωμένοι στο σεβασμό του χάρτη. Η γνωμοδότηση που μας έχει παρουσιαστεί φαίνεται να είναι πολύ ε, ισορροπημένη, βασίζεται στις αρχές της συνθήκης. Υπάρχουν κάποια ζητήματα μόνο τα οποία θέλει η Μπάρμπαρα να συζητήσει διμερώς με τον συγητή. Το ΕΛΚ θα υποβάλει τροπολογίες προκειμένου η γνωμοδότηση να καταστεί πιο ισορροπημένη και να προβλέπει κάποιες, κάποιες συγκεκριμένους κανόνες ε, επίσης έχουμε κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά την αιρεσιμότητα για τα ευρωπαϊκά δικαιώματα υπό ε, το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όλα αυτά βεβαίως θα αντικατοπτρίζονται και στις τροπολογίες μας. Ευχαριστώ. Ε, λέει ο Πρόεδρος. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει το λόγο. Θέλεις να αντικαταστήσεις την ε, κυρία Μπόνφροϊ, την ισχυώδη συγγύτρια των σοσιαλιστών. Ναι. Αυτό θέλω να κάνω και θέλω να ζητήσω συγγνώμη που η Κριστίν δεν ήταν εδώ, δεν είναι εδώ, λόγω μια ξαφνική συνάντηση που είχε στο Παρίσι. Θα σα διαβάσω τι τις σημειώσεις της. Τι λέει η Κριστίν, θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον εισηγητή, τον κύριο Ντεγιόν, για τι εξαιρετικέ του προσπάθειες. Συμφωνώ με τα οικονομικά και κοινωνικά θέματα που υπογραμμίζει. Δεν δίνεται επαρκή προσοχή στι κοινωνικέ διατάξει του χάρτη όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση τη Ένωση παρότι επηρεάζουν τα κοινωνικά δικαιώματα που θεσπίζονται στο χάρτη όπως η παιδεία και η κοινωνική ασφάλεια που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Υποστηρίζω επίσης το αίτημά του για επιτάκυνση των διαπραγματεύσεων για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εγώ θα υποβάλω με στις επόμενες ημέρες κάποιες τροπολογίες με εστίαση την υλοποίηση του χάρτη από τα κράτη-μέλη. Το άρθρο 51 αναφέρει ότι ο χάρτης ε, εφαρμόζεται μόνο κατά την υλοποίηση, κατά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Αλλά πολλές αποφάσεις και η πολυάριθμη νομολογία έχουν δημιουργήσει σύγχυση. Χρειαζόμαστε διευκρίνηση του άρθρου αυτού που σε τελική ανάλυση βοηθά τα κράτη-μέλη για καλύτερη υλοποίηση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάτι τελευταίο. Θεωρώ και εγώ ότι είναι θετική επιρροή του χάρτη μας επιτρέπει προενεργά μέτρα προστασίας ε, και διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι πολύ σημαντικό να δράσουμε γρήγορα, να δράμε μόλις αισθανόμαστε απειλή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το θέμα είναι τεχνικό, παρόλα αυτά δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία να στείλουμε ένα χειρό πολιτικό μήνυμα σε ε, μια συνέντευξη στο Λουξεμβούργο πριν μερικέ εβδομάδε ε, υπουργών δικαιοσύνη. Η Πολωνία μπλόκαρε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη για πρώτη φορά. Είναι άνευ προηγουμένου αυτό. Ο χάρτης μας και οι βασικές μας αρχές βρίσκονται ε, υπό επίθεση. Γι' αυτό εγώ θα συνεργαστώ με τους ηγητές και τους ε, Ευχαριστώ. Έχουμε κλείσει. Τι κύριε Διόγκ, έχετε άλλα λόγια, όχι. Κοιτάξτε, εν συντομία, ε, αναμένω να δω τις τροπολογίες ε, η προθεσμία δεν ξέρω την έχουμε. Νομίζω ότι είναι σύντομα σχετικά. Δεν τη βρίσκω τώρα. 12 Νοεμβρίου λέει ο πρόεδρο. 12 Νοεμβρίου, 5 η ώρα το απόγευμα. Δική μου δουλειά είναι να σα το πω. Λέει ο πρόεδρο. Γι' αυτό με πληρώνω όλα αυτά τα ε, σεβαστά ποσά για να το λέω αυτό στο τέλος. 12 Νοεμβρίου, 5 το απόγευμα. Είμαι ευγνώμων, καθώς φτάνουμε στο τέλος ε, της εντολής ε, του Κοινοβουλίου, της θητείας του Κοινοβουλίου όλο και περισσότερα μέλη λείπουν, αλλά εξακολουθεί σκληρή δουλειά από τους συντονιστές, από τα μέλη που έρχονται και αναγνω... αναγυγνώσκουν τις δηλώσεις τους. Αλλιώς δεν θα κάναμε δουλειά. Ευχαριστώ και το προσωπικό για όλα τα σημειώματα που συντάσσει. μα βοηθά πάρα πολύ. αλλιώ, δεν θα δίναμε απαντήσει στα σχέδια όλα αυτά γνωμοδοτήσεων και εκθέσεων. Θέλετε, είπατε από την Κομισιόν. Μπάρμπαρα Νόλαν από την Κομισιόν εδώ. Θέλετε να μιλήσετε γι' αυτό, Μπάρμπαρα. Έχετε το λόγο αν θέλετε. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλωσορίζουμε και εμείς αυτή τη γνωμοδότηση και συγχαίρουμε τον κύριο Ντεγιόγκ, τον εισηγητή. Και εμεί ε, τον ίδιο στόχο έχουμε μεγαλύτερη προβολή, μεγαλύτερη εφαρμογή, καλύτερη χρήση του χάρτη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα ευρωπαϊκά όργανα και από τα κρατημέλη και από την κοινωνία των πολιτών. Απλά να πω ότι παρατηρείται μια κινητικότητα όσον αφορά τη σύμβαση. Και πάλι έγιναν συζητήσεις στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου, παρατηρείται λοιπόν κάποια κινητικότητα που θα οδηγήσει πιστεύουμε σε κάποια πρόοδο στο ζήτημα αυτό και αυτή είναι καλή είδηση για πριν κλείσουμε σήμερα. Αναμένουμε να δούμε την επόμενη εξέλιξη της ε, γνωμοδότησης. Ευχαριστούμε Μπάρμπαρα, ευχαριστούμε που ήρθατε και πάλι εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε κύριε Ντεγιόνγκ για τη γνωμοδότηση. Προθεσμία 12 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ συνάδελφοι προτείνω να κάνουμε διάλειμμα μέχρι τις 5 και 45, 6 παρατέταρτο, όπου θα ξεκινήσει η ψηφοφορία. Κάνουμε διάλειμμα μέχρι εκείνη την ώρα. Ευχαριστώ. Σε τρία λεπτά, συνάδελφοι, ε, πάρτε τις ε, κάρτες σας για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Oh, sorry. <laughs> Don't need to give anyone a, a shock. Uh, colleagues, uh, we uh, beginning. Λοιπόν, συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Ανεξαρτήτως του ποιος είναι εδώ, γιατί έχουμε πολλές ψηφοφορίες. Τέσσερις, συν μία για, την, για τον οργανισμό επιτήρησης. Έχουμε αρκετές μακροσκελεί ψηφοφορίε ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων για το μήκος τη διαδικασία. Θα γίνουν και σήμερα και την Πέμπτη, αλλά μία από τις μεγάλες ομάδες δεν θα είναι παρούσα την Πέμπτη και επομένω, και πάλι στο συγγνώμη εκ των προτέρων για το μακροσκελές αν συγκεντρωθούμε ίσως να τα καταφέρουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και τα καλά νέα είναι ότι δεν θα έχουμε και τόσα πολλά Στρασβούργο την ερχόμενη εβδομάδα. Τόσο μάλλον τα σχετικά καλά νέα. Γιατί έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μέχρι το τέλος εντολής. Ξεκινώ αμέσω με την πρώτη. Η συγκέντρια δεν είναι εδώ. Αλλά είχαμε και την γνωμοδότηση ΛΥΜΠΕ για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που αντικαθιστά το ισχύον. Ο φάκελος εδώ έπρεπε να ε, προχωρήσει γρήγορα λόγω των προθεσμίων και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις για την συλλογική τους προσφάρια. Προσπάθεια δεν είναι εδώ η συγγήτρια αλλά είναι εδώ η σκιώδης. Κάποιος μου κάνει νόημα από ό,τι φαίνεται. Ναι πρόεδρε. Εγώ έφτασα χωρίς κάρτα και θα ήθελα να μπορέσω να ψηφίσω διανάτα τη χειρός, αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε. Καθότι έχετε την πιο προβληματική από τέσσερις ψηφοφορίες. Ίσως κάποιος θα μπορούσε να σας φέρει μια κάρτα και στο μεταξύ θα καταγράφουμε βέβαια την ψήφο σας. Μέχρι να φτάσουμε σε εκείνη την ε, ε, ελπίζω να ελέγξετε όλοι ότι έχετε την ηλεκτρονική κάρτα σας. Εν πάση Είναι κανένα άλλος. Όχι. Ωραία. Άρα τις έχετε όλοι. Έλεγα λοιπόν ότι πάμε τώρα στην ψηφοφορία για την ε, πρόταση κανονισμού για το Social Fund Plus. Συμβαστική 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 121 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 16. Πέρας. Εγκρίνεται. 133. Άρχεται η ψηφοφορία. Όχι. Όχι, λέει ο πρόεδρος. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Συμβαστική 17, παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 18. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 19 παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 20 παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 21. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 22. Παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 23. Παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 24 παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 25. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 26. Πέρας. Εγκρίνεται. 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 161 τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 27. Παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 165, παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 166. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 28, παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 171, παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 172. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 29, παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται.

Πέρας. Εγκρίνεται. 180 άρχη της Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 30 παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 31 Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβεσ... Τροπολογία 185. Παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 186. Πέρας. Εγκρίνεται. 187. Πέρας Εγκρίνεται 188. Πέρας. Εγκρίνεται 189. Πέρας. Απορρίπτεται. 43 παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 32. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 45. Πέρας. Εγκρίνεται. 191 παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται 192. Πέρας. Εγκρίνεται 193. Πέρας. Εγκρίνεται 194. Πέρας. Εγκρίνεται 46. Πέρας. Εγκρίνεται 47. Πέρας. Εγκρίνεται. 195. Πέρας. Απορρίπτεται. 196 παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 48 τροπολογία. Πέρας εγκρίνεται 49 πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 33. Παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 51 τροπολογία. Πέρας. Εγκρίνεται 52. Πέρας εγκρίνεται 198 πέρας απορρίπτεται πάμε στα παραρτήματα 199 τροπολογία πέρας απορρίπτεται από κοινού 200 και 201 παρακαλώ πέρας απορρίπτονται 53 και 54 πέρας εγκρίνονται 203 παρακαλώ πέρας εγκρίνεται από κοινού 55 και 56 παρακαλώ πέρας Εγκρίνονται. 204 και 205 παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτονται. Από κοινού 57 και 58. Πέρας. Εγκρίνονται. Από κοινού 206 και 207 παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται. 59 παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 60. Πέρας. Εγκρίνεται αιτιολογικές 61 τροπολογία. Πέρας. Εγκρίνεται 62. Πέρας. Απορρίπτεται 63. Πέρας. Απορρίπτεται. 64. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1, παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 70. Πέρας. Απορρίπτεται. 69. Πέρας. Απορρίπτεται. 71 και 72 είναι ταυτόσιμες παρακαλώ. Και 2. Πέρας εγκρίνονται. Συμβαστική 2. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 παρακαλώ. Πέρας. 81 παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Η παριθμόν είναι 6. Πέρας. Εγκρίνεται. 83. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Υπαριθμό 89 τροπολογία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7α. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 99. Πέρας εγκρίνεται 101 πέρας απορρίπτεται 102 πέρας εγκρίνεται 9 πέρας εγκρίνεται. Συμβαστική 8 πέρας εγκρίνεται. Συμβαστική 9 πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 106 πέρας εγκρίνεται. Συμβαστική 10 πέρας εγκρίνεται 109 πέρας εγκρίνεται συμβαστική 11 παρακαλώ πέρας εγκρίνεται αυτές μπορούμε από κοινού να τις ψηφίσουμε όχι δεν μπορούμε δεν μπορούμε αλλά προσπάθησα 114 λοιπόν τροπολογία Πέρας. Εγκρίνεται 115. Πέρας. Εγκρίνεται 14. Πέρας. Εγκρίνεται 15. Πέρας. Εγκρίνεται 16. Πέρας. Εγκρίνεται. 116. Πέρας. Εγκρίνεται. 117. Πέρας. Εγκρίνεται. 17. Πέρας. Εγκρίνεται. 118. Πέρας. εγκρίνεται 18. Πέρασε. Λοιπόν, ονομαστική, παρακαλώ. Πέρασε. Εγκρίνεται 31 υπέρ 7 κατά καμία εποχή. Πάμε απευθεία στην επόμενη. Αν θέλει κάποιο ένα διάλειμμα να μου το πείτε, αλλιώ προχωρώ απευθεία. Πάμε στη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027. Η συγκεκριτή είναι ο Γερούν Λέναρς. Θέλετε το λόγο πριν από την ψηφοφορία. Όχι, όπως υποψιαζόμουν. Πάμε στην τροπολογία 63. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ψήφισαν άπαντες. Ζητώ συγγνώμη συναδελφοί. Ξαναδιαβάζω, μιλάμε για την έκθεση του κύριου Λενάρς. Ξεκινάμε με την τροπολογία 63, Άρχιτε ψηφοφορία. Το ξανακάνουμε για λόγους που δεν κατάλαβα καλά. Πέρας εγκρίνεται. 64. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 14 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 15 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 16. Πέρας. Εγκρίνεται. 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται 66 άρχεται ψηφοφορία 68 συγγνώμη πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται συμβιβαστική 9 άρχεται ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται τροπολογία 74 άρχεται ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10α έρχεται ψηφοφορία. 10α. Πέρας. Εγκρίνεται. 10b. Συμβιβαστική όχι καταπίπτει. Πάμε στη συμβιβαστική 11α. 11α έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11β. Συγγνώμη. Καταπίπτει. Πάμε στην τροπολογία 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 27. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 93. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 94. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη. 95. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. 96 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 97 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 98 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 99 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 100 άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 101 άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις 29. Τροπολογία άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται 1 άρχιτη ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται συμβιβαστική 1 άρχιτη ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται συμβιβαστική 2α άρχιτη ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται συμβιβαστική η τροπολογία, συγγνώμη, 36 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 37 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 38 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 4, συμβιβαστική, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 43, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 44. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 45. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 46. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 47. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 48. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 49. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 50. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 7. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική, ε, συγγνώμη, τροπολογία 54, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 55, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 56, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται συμβιβαστική 6, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 59. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 61. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται Ονομαστική ψηφοφορία. Τέλος, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 34 υπέρ, 1 κατά και 4 αποχές. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και πάμε απευθείας στην επόμενη ψηφοφορία πλήρης εφαρμογή του και εκτιμένου του Σέγγεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Κύριε Στάνισεφ, θέλετε το λόγο. Ωραία, περνάμε στην ψηφοφορία. Περνάμε στην τροπολογία 17. Amendment 17, the vote is now closed. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται και αυτή. Τροπολογία 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 9. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται και αυτή. Συμβαστική 11. Ψηφίστε παρακαλώ. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 36. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 37. 39, με συγχωρείτε. Συγγνώμη, συγγνώμη. 39, ψηφίστε παρακαλώ, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 12. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15. Άρχεται ψηφοφορία. Επί της τροπολογίας, της συμβαστικής τροπολογίας 15. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Επίσης εγκρίνεται. Πάμε στις αιτιολογικές αναφορές. Συμβαστική 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ετολογικές σκέψεις. Συμβαστική 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται επίση και τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία ψηφίστε παρακαλώ μπράβο Σέργη και Άννας πολύ ωραίοι συμβιβασμοί γρήγορα τελείωσαν την ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 36 υπέρ 4 κατά και μια εποχή. συγχαρητήρια στον εισηγητή και μπράβο του λοιπόν και μιας και ανεφέρθηκα σε μακροσκελείς ψηφοφορίες που θα έχουμε, περνάμε στην τέταρτη και τελευταία ψηφοφορία πριν περάσουμε στο προσωπικό του Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών. Εδώ μιλάμε για μια γνωμοδότηση για την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του εθνοσιακού δικαίου που θα ψηφιστεί από την Επιτροπή Γιούρη τον Νοέμβριο έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα σε κάποιε από τι προτα... Ε, ε, διατάξει τη πρόταση, ιδίω όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επίση, έχουμε κοινή αρμοδιότητα σε κάποια άλλα ζητήματα, όπω είναι τα, ε, οι, οι ποινικέ υποθέσει που σχετίζονται με του ε, πληροφοριοδότε. Συντάκτρια τη γνωμοδότηση είναι η κυρία Ρουή. Αν θέλει τον λόγο, όχι, δεν τον θέλει. Ωραία, άρα μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στην πληροφορία. Να σα προειδοποιήσω συνάδελφοι ότι δεν έχουμε πολλούς συμβιβασμούς, γι' αυτό και χρειάζεται πειθαρχία από όλους. Τροπολογία 33. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 166. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 175. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 176. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 177. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με μικρή διαφορά. 179. Ψηφίστε παρακαλώ. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Εγκρίνεται. 180. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 181. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική 3. Άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 191. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 192. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 193. Άρχιτε η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 194 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 199. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 200. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 201. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 203. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 208. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 211-212 που ταυτίζονται. Αρχίστε, ψηφίστε παρακαλώ. Εγκρίνεται. 213. Άρχισε η ψηφοφορία. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Εγκρίνεται. 214-215 που ταυτίζονται. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέραστης τη ψηφοφορία. Εγκρίνονται. 216. Ψηφίστε παρακαλώ. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Απορρίπτεται. 221. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Παρακαλώ. Πέρας Εγκρίνεται. 2.28 τροπολογία. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.29. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7. Ναι, όχι, πρέπει να κάνουμε την 230 πριν την συμβαστική 7. 2.30 λοιπόν, ακυρώνω τη συμβαστική 7 την ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 2.30 τροπολογία παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα μπορούμε να ψηφίσουμε τη συμβαστική 7 και ζητώ συγγνώμη. Συμβαστική 7. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2.33. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.34. Θα πάω λίγο πιο αργά γιατί βλέπω ότι έχουμε οριακέ πλειοψηφίε. Πάντω αυτή εγκρίνεται. 2.35. Όχι και πολύ αργότερα, μην ανησυχείτε. Πέρα. Εγκρίνεται 2.36. Πέρας, εγκρίνεται 2.39. Πέρας, Εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 242. Πέρας. Απορρίπτεται 243. Πέρας. Απορρίπτεται 2.44 πέρας απορρίπτεται 2.48 πέρας εγκρίνεται 2.49 και 2.50 ταυτόσιμες παρακαλώ πέρας εγκρίνονται. 2.51 πέρας. Εγκρίνεται. 2.52 πέρας. Εγκρίνεται. 2.54 πέρας Εγκρίνεται 2.55. Πέρας. Εγκρίνεται 2.56. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 261. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.64. Όχι, ζητώ συγγνώμη, 2.63. 2.63. Αρχή τη ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 2.64. Πέρας. εγκρίνεται 265 πέρας εγκρίνεται 266 πέρας εγκρίνεται 267 όχι 268 268 πέρασε εγκρίνεται συμβαστική 11 Πέρας. εγκρίνεται, 2,71. Την έκανα την 11 λέει ο πρόεδρος. Μόλις την έκανε. 2,71. Πέρας. Εγκρίνεται. 2,73. Πέρας. Εγκρίνεται. 2,76. Πέρας. Εγκρίνεται. 2,78. Πέρας. Απορρίπτεται. 2,99 Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 12. Όχι και πάλι το συγγνώμη πρέπει πρώτα να κάνουμε την τροπολογία 280 παρακαλώ. Το μηχάνημα έτσι αλλιώς δεν δούλευε. 280. Ήξερε το μηχάνημα λέει ο πρόεδρος. Τώρα πέρασε για τη 280. Ίσως να κουράζεται και να έχει κουραστεί και το μηχάνημα λέει ο πρόεδρος. Και λέμε, λέει ο πρόεδρος του σχολή που δεν ακούσαμε, μη μου το λέτε αυτό. Απορρίπτεται πάντως η 280. Και συντός συγγνώμη Μπάρμπαρα. Um, λοιπόν, συνάδελφοι, συμπαθάτε με, αλλά έκανα κι άλλο ένα λάθος. Δεν ψηφίσαμε τη 267. Μα δεν την ψηφίσαμε. Δεν ψήφισα την 267 πριν τη συμβαστική 11, λέει ο πρόεδρος. Sorry, Ας παρακαλώ να ψηφίσουμε τη 267, παρακαλώ. Πέρασε. Εγκρίνεται. Άρα επανερχόμαι τώρα στη συμβαστική 12. Συμβαστική 12 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 285. 285, έτσι. Πέρας. Απορρίπτεται. 287. Όχι, όχι, όχι, ούτε τώρα. Πρώτα η 286. Η 286, ναι. Ναι, 286 ψηφίζουμε παρακαλώ. 286. Πέραστε για, το, για τη 286. Ψηφίσατε τη 286 όλοι, λέει ο πρόεδρος ενώ έχει κλείσει η ψηφοφορία. Right. everyone voted? Άρα το ερώτημα απευθυνόταν σε όλους συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου. Εγκρίνεται με μία ψήφο, μια και ψήφισε και ο πρόεδρος επιτελούς την 286 και ευχαριστώ το συντονιστή είναι η πρώτη ενδιαφέρουσα ζήτηση που είχαμε όλη τη βδομάδα. 2.87. Και ζητήσω συγγνώμη και πάλι λέει ο πρόεδρος, κουράζομαι τώρα σιγά σιγά και εγώ 2.87 παρακαλώ. Yeah, no, no, I know. The vote is closed. Πέρας ε, της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Δύο, και 22 ταυτόσιμες άρχεται η ψηφοφορία. Έχασα τη φόρα μου. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.91. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.92. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται συμβιβαστική 14. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται συμβιβαστική 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 308 τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρινεται 3.11 3-11 άρχεται ψήφισαν απαντές πέρας για όνομα του Θεού η ομάδα μου λέει ο πρόεδρος απορρίπτεται ε, πέρας ψηφοφορίας Oh God. Um, look, we have to now vote all these. Συγγνώμη, πρέπει να ψηφίσουμε τώρα όλε τι άλλε ε, διότι δεν είμαι βέβαιο τι έγινε. Να ελέγξουμε την 3.11 πριν. Γιατί αλλιώς, ε, ε, κοίταξε, το μόνο που λέω, έχουμε άλλε 15 εκατομμύρια ψηφοφορίε εξαιτία αυτό Τι με νοιάζει εμένα η αρχή. Έχουμε ένα κάρο ψηφοφορίες. Δεν ξέρω εσεί αλλά εγώ είμαι λίγο κουρασμένος. Εντάξει, εντάξει. 3.12 λοιπόν την ψηφίσαμε. 3-12 ψηφίζουμε τώρα. Προσπαθώ. 3-12. Άρχεται η ψηφοφορία. Τι με νοιάζει αρχή. Απλά το λέω έτσι για να... Πέρας. Εγκρίνεται, συγγνώμη. 3-13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 3-14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 3.15 άρχεται. Πέρας. Να... Ε, απορρίπτεται. 3.16 άρχεται η ψηφοφορία πέρας. Απορρίπτεται πιθανότατα. Απορρίπτεται. 3.17 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 318 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 319 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 320 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 321. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 326. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στην 341. 341 δείξαμε μια ολόκληρη σελίδα. 3.41. 3.41. Ψήφισαν άπαντες, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 3.46 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 347 αρχή ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται συμβιβαστική 17 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 350 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 3.53. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 3.55. Άρχεται η ψηφοφορία. Είναι μικρή η διαφορά πλειοψηφίες, οπότε μας προσέχουμε. 3.55 πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 356 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας απορρίπτεται. 357 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας απορρίπτεται. Συμβιβαστική 18 άρχεται η ψηφοφορία. Συμβιβαστική 18. Θέλετε να βάλετε την κάρτα σας. Δουλεύει. Ψηφίστε την συμβιβαστική 18. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 361. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 362. Άρχεται η ψηφοφορία. Ποιος είπε όχι. Πέρας. «362, ναι. Ποιος είπε όχι, γιατί λέτε όχι. 362 είναι. Να είπατε ναι. Α, εντάξει. Πέρας ψηφοφορίας. Συγγνώμη, εγώ δεν ψήφισα. Πέρας. Εγκρίνεται. 364. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 365. Άρχεται η ψηφοφορία. Μόνικα, δεν ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 366. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 367. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 368. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 369. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται συμβι... 3, 80 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Πέρας. Απορρίπτεται 22 συμβαστική άρχεται ψηφοφορία. Συμβαστική 22 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Όλα είναι εντάξει. Όλα εντάξει. 383. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 384 η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 385 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 386 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Πέρας. Εγκρίνεται. 387 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Κάνεις πλάκα, λέει ο πρόεδρος στην συνάδελφό του. Η Σουηδία 381 ψηφίσατε. Λοιπόν, 381 δεν ψηφίσαμε. Πάμε γρήγορα στην 381. Ζητάω συγγνώμη, συναδελφοί. Πηγαίνετε πάνω πίσω στην 381. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας απορρίπτεται. Πάμε ξανά προς τα κάτω στην 388. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Επιλογές αναφορές 34 ε, ε, πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 35 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Πέρας. Εγκρίνεται. 36 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται επίσης 37 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 38. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται συμβαστική 23. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται τροπολογία 44. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται τροπολογία 45. αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται συμβεστική 24. αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 52. αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 53, έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβεβαστική 25, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 57. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 58. Η... Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται συμβιβαστική 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται 62 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 63 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 64 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 66 άρχεται ψηφοφορία. Συγγνώμη, 65 άρχεται ψηφοφορία. 65. Πέρας. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 66 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 68. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 70. Άρχεται η ψηφοφορία. Συγγνώμη. 69. 69 είναι. Ε, Δεν είχα δίκιο. 70. Δεν είχα δίκιο. 70 λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεν είχα δίκιο. 69. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Και τώρα πάμε στην 70. Όχι στην 5. 5. Τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 70 η αγαπημένη μου άρχιτη ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 71 άρχιτη ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 27 άρχιτη ψηφοφορία Συμβαστική 27 πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις, τροπολογία 6 Α, ε, πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 28 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 29 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Έγκρινεται συμβαστική 30, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται η συμβαστική 31, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται τροπολογία 83, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 84, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 85, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 86, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 9, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 88 έρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 89 έρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 91 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 93. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 97. Άρχεται ψηφοφορία. Όχι. Καταπίπτει. Συγγνώμη. 94. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ε, 95. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 96. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Αφήνουμε την 96, δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε. Πάμε στην 97. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 98. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασική 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 99. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 102. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 103. άρχισε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 104. Άρχιστη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 106. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 33. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 113. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 114. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 115. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 13. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 116. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 35. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 120 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 121 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 122 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. 123 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 124 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ωραία μουσική. 125 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον αυτό το ringtone. Μ' αρέσει. Λοιπόν, πέρας της ψηφοφορίας επί της τροπολογίας 125. Όχ, τι έπαθε αυτό το μηχάνημα. Χάλασε. Παναγιά μου. Πάμε ξανά, 125. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 126 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 128. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 129. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 130. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 131. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 132. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίπτεται. 133. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίνεται. 134. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 135. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 136. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 137. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 138. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. 139 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 140 ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίνεται. 141 ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 142 ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 143. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 144. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. 145. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 147. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 148. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 149. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίπτεται. 150. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Rejected. 152. votes, 151. 151. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 152. Ω, συγγνώμη, εγκρίνεται, εγκρίνεται. 152. Ψηφίστε παρακαλώ. Εγκρίνεται. 153. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 154. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 155. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 159. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Εγκρίνεται. 26 υπέρ, 8 κατά, 4 εποχές. Συγχαρητήρια στον συγκητή. Λοιπόν, συνάδελφοι, έχουμε μία τελευταία γρήγορη ψηφοφορία. Έχουμε τρεις υποψήφιους για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τοξικομανίας και Ναρκωτικών. Θα το κάνουμε πολύ γρήγορα. Στην ουσία ψηφίζεται θα πάρουμε κάθε υποψήφιο. Συνάδελφοι, ακούστε μου λίγο σας παρακαλώ, για να μπορέσουμε να φύγουμε. Λοιπόν, ξαναλέω. Θα αναφέρω τους τρεις υποψήφιους και θέλουμε δύο για το κέντρο. Αυτός που θα χάσει, που θα έχει τις λιγότερες ψήφους, θα είναι ο αναπληρωματικός. Θα πω τα τρία ονόματα. Όταν θα λέω το όνομά του, πατήστε το πράσινο κουμπί, αν τον θέλετε, αυτόν τον υποψήφιο. Μην κάνετε τίποτα άλλο. Απλά περιμένετε να ακούσετε το όνομα του υποψηφίου που θέλετε. Αν, αν πατήσετε ε, το κόκκινο ή την αποχή δεν θα προσμετρηθεί έτσι κι αλλιώς. Ψηφίζετε με το πράσινο κουμπί καταφατικά ε, υπέρ του υποψηφίου που θέλετε. Θα σας πω τα τρία ονόματα και θα καταγραφούν μόνο οι θετικές ψήφοι. Αυτά εν συντομία, είχα και πολύ περισσότερα να πω, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Ε, έμαθα και το ex aequo μια λατινική ορολογία, έναν λατινικό όρο που δεν τον ήξερα. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Υπήρχαν και πολλά άλλα να πω, απλά θα σας τσάτιζα όμως, γι' αυτό σας λέω το βασικό, το ζουμί. Ψηφίστε υπέρ του υποψηφίου που επιθυμείτε. Εντάξει, όχι και πολύ μυστική η ψηφοφορία. Εν πάση περιπτώσει, κάντε το έτσι όπως σα το λέω για να τελειώνουμε. Λοιπόν, πάμε. Wolfgang Goals. Gertz. Συγγνώμη. Μπορείτε και να απόσχετε από την ψηφοφορία άμα αυτό θέλετε να κάνετε. Δεν θα σα το απαγορεύσει κανείς. Έλλη Μαλιόρη. Α, ναι, συγγνώμη, η προηγούμενη ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. 27 ψήφοι υπέρ του υποψηφίου αυτού. Νέλη Μαριόρη. Ποιος προκρίνει αυτήν την υποψήφια. Okay, we're now on Maliori. So if you want to vote for Maliori, vote positively. If you don't want... Αν θέλετε τον συγκεκριμένο υποψήφιο, ψηφίστε υπέρ του. Αν δεν τον θέλετε, μην κάνετε τίποτα. Μπορείτε να ψηφίσετε και κατά, αλλά δεν θα προσμετρηθεί η ψήφο κατά. Λοιπόν, υπήρξε κάποιο μπέρδεμα με τον πρώτο. Ωραία. Να το ξαναπώ. Είναι αυτοί οι υποψήφοι για τον οργανισμό. Μπορείτε να κάνετε λίγο ησυχία σας παρακαλώ για να μην γίνουν λάθη, επειδή είμαστε και κουρασμένοι, να ξαναρχίσουμε από την αρχή. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Όταν θα λέω το όνομα, ακούστε προσεκτικά, όταν θα λέω το όνομα του υποψηφίου, αν τον θέλετε αυτόν τον υποψήφιο, αν θέλετε να τον υπερψηφίσετε, ψηφίστε με το πράσινο κουμπί. Άμα δεν θέλετε να ξέρουν οι άλλοι τι ψηφίζετε, ψηφίστε αποχή. Έτσι και αλλιώς οι αποχές και οι ψήφοι κατά δεν θα προσμετρηθούν. Άμα θέλετε να είναι μυστική η ψηφοφορία, μπορείτε απλά να πατήσετε αποχή για να μην ξέρει κανεί τι έχετε ψηφίσει. Έχετε βάλει το χέρι σα στο μηχάνημα, αλλά δεν ξέρουμε τι ψηφίζετε. Και όλε οι θετικέ ψήφοι θα προσμετρηθούν στο τέλο. Όλε οι άλλε ψήφοι απλά δεν θα συνυπολογιστούν. Εγώ στο, θα λέω τα ονόματα και θα καταγράφονται μόνο οι θετικέ ψήφοι υπέρ του κάθε υποψηφίου. Wolfgang, ψηφίστε για τον Wolfgang, παρακαλώ. Gertz. Ψηφίζουμε υπέρ του Wolfgang Goetz. Όποιος θέλει να τον ψηφίσει, ας τον ψηφίσει τώρα. Λοιπόν, τώρα έχουμε 19 θετικές, 7 κατά 8 αποχές. Οι 19 είναι αυτές που μας ενδιαφέρουν. Νέλη Μαλιόρη. Ψηφίστε παρακαλώ. So, The vote is still open. The vote is now closed on many Maliori. And... Πέρας της ψηφοφορίας, Μαλιόρι πήρε 30 ψήφους και τρεις κατά τέσσερα δεν μας νοιάζει κιόλας. Και μετά Σαμπράντσκι. Ψηφίστε παρακαλώ για τον Σαμπράντσκι, τον ή την. Δεν διευκρινίζει ο Πρόεδρος. Πέρας. Εδώ έχουμε 18 ψήφους υπέρ. Οπότε, Γκέτς και Μαλιόρι είναι τα τακτικά μέλη και Σαμπράνσκι είναι ο αναπληρωματικός. Ανεσυγγνώμη, ναι, να κάνουμε μια τελευταία τελική ψηφοφορία. Δεν ξέρω γιατί, αλλά για τη διαδικασία χρειάζεται να γίνει και μια τελική ψηφοφορία για όλα τα επιλέξιμα μέλη και να επιτευχθεί και απόλυτη πλειοψηφία. Πώς ψηφίζουμε κανονικά, έτσι. Βάλτε το δαχτυλάκι σας, ψηφίστε για να... ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά. Ψηφίστε στο μηχάνημα ποιος είναι υπέρ αυτού του καταλόγου υποψηφίων, έτσι όπως καταρτίστηκε. Ωραία, έχουμε απόλυτη πλειοψηφία, μπορείτε να φύγετε, σας ευχαριστώ, γεια σας. Ολοκληρώσαμε τι ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ για την υπομονή. Ευχαριστώ για όλα. Γεια σας συνάδελφοι. Ήταν πολύ μακροσκελής η ψηφοφορία αυτή. Αλλά εντάξει, τα καταφέραμε. Καλό βράδυ.